και, η Τσεχία είναι μέλος της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την Πολωνία. Πράγματι αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς είπα και εγώ όταν ευχαρίστησα τους κυρίους Ντόλ και Σούλτς για την ε, συνεισφορά τους και σας ευχαριστώ και σας κύριε Μπεζίνα που το επισημάνατε πράγματι είναι καταστροφικές οι πλημμύρες. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην ημέρια διάταξη. Έχουμε την απλοποιημένη διαδικασία για την έκθεση του κυρίου Γκρέχ σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Μία μονάχα ψηφοφορία υπάρχει με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. <clears throat> Πέρα της ψηφοφορίας. «578 ψήφοι υπέρ, γίνεται δεκτή η έκθεση. Στη συνέχεια έχουμε πάλι με απλοποιημένη διαδικασία την έκθεση Schmidt για τον διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, μια νέα εταιρική σχέση στην Ευρώπη. Μία μονάχα ψηφοφορία. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η ψηφοφορία στην έκθεση της κυρίας Χάρμς για την οικονομική υποστήριξη σε ό,τι αφορά την θέση αχρηστία των ε, αντιδραστήρων 1 και 4 του Κοσλοντού στη Βουλγαρία. Ψηφίζουμε λοιπόν για τις τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής, αμπλόκ μαζί, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Έχουμε τώρα τις μεμονωμένες ψηφοφορίες, τροπολογία 6 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Επίσης 10 από την Αρμόδια Επιτροπή ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 1, έχουμε δύο τροπολογίε. Την 35 των Πρασίνων έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 21 της Αρμόδιας Επιτροπής Βιομηχανίας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 2, τροπολογία 36 των Πρασίνων, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Δεν γίνεται δεκτή η τροπολογία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 22 της Αρμόδιας Επιτροπής. Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το, την αιτιολογική σκέψη 6 έχουμε τροπολογία 32 των πρασίνων ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 της Επιτροπής Βιομηχανίας ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 33 των πρασίνων με ονομαστική ηλεκτρονική. Θέλετε έλεγχο για την 7. Εντάξει, ελέγχουμε την 7 πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία ελέγχου. Για την 7 της Επιτροπής βιομηχανία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Πράγματι και de facto εγκρίνεται. Τροπολογία 33 των Πρασίνων ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη <clears throat> Δεν γίνεται δεκτή η τροπολογία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 8 της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Μετά την αιτιολογική σκέψη 13 έχουμε δύο τροπολογίες. Πρώτα τη 34 των Πρασίνων. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. <clears throat> Έλεγχος για την τροπολογία 34 Αρχίεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται λοιπόν. Πραγματικά. Τροπολογία 20 αρμόδιας επιτροπής. Ψήφι Κατά αποχές δεκτή. Το ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Δεκτή. Δεκτό το ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική και πάλι κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Δεκτό το ψήφισμα. Ακολουθούμε, ακολουθεί η έκθεση Φανής Λερόι για τις συνεργίες μεταξύ της ε, ε, έρευνας και της καινοτομίας. Ο εισηγητής έχει ζητήσει να λάβει το λόγο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θέλω να ζητήσω ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ ονόματος του ΕΛΚ. Έχει περάσει η προθεσμία, αλλά αν δεν έχει κάνει αντίρρηση, τότε νομίζω δεδομένων των περιορισμένων δυνατοτήτων που είχαμε αυτή την εβδομάδα προτείνω να έγινε κάτι τέτοιο. Έχει κάποιο αντίρρηση, όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε ονομαστικά την έκθεση Φάνη Στελοϊάρχη τη ψηφοφορία. Die Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Κατόπιν έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση Χουανγκόκ για τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψη. Έχουμε πολλές ονομαστικές ψηφοφορίες. Τροπολογία 1, όπως αναθεωρηθήκε, ή 1 έως 11 έχουν αναθεωρηθεί. Λοιπόν, τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία και να σας ανακοινώσω πως ζητήθηκε να μην ψηφίσουμε ένα μπλοκ. Λοιπόν, τροπολογία 2 άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. αρχιτή η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας λοιπόν. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 7, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 8, Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην παράγραφο 2. Ψηφίζουμε για το αρχικό κείμενο σε χωριστή ψηφοφορία. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτό παράγραφος 4 το αρχικό κείμενο σε τρία μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται μέρος τρίτο υπέρ θέλετε να επαληθεύσουμε το, μέλος, το μέρος δεύτερον άρχιτη ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται τρίτο μέρος υπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφος 7. Το αρχικό κείμενο. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Ψηφίζουμε την παράγραφο 11, το αρχικό κείμενο, πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό παραγραφος 17 το αρχικό κείμενο σε τρία μέρη μέρος πρέπει να σας πω πως κάποιες ε, ονομαστικές ε, ψηφοφορίες ε, αποσύρονται μέχρι την τελική ψηφοφορία. Πρώτο μέρος λοιπόν της παραγράφου 17 υπέρ, κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος τρίτο υπέρ, κατά. Αποχές θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 19, τροπολογίο 9 του εισηγητή, όπως άλλαξε. Με συγχωρείτε, δεν έχει αποσυρθεί αυτή η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην παράγραφο 19 του αρχικού κειμένου. σχολιστή ψηφοφορία, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά άποχες θα το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία. Μέλος, μέρος δεύτερο της παραγράφου 19 του αρχικού κειμένου. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 59, το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, με συγχωρείτε. Γίνεται δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Δεκτό. Παράγραφος 61. Το αρχικό κείμενο ψηφίζουμε σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος περ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο μέρος περ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται εκτιμώντας α σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές. Και αυτό γίνεται δεκτό. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. γίνεται δεκτό με 302 έναντι 275 ψήφων. Ο εισηγητής ζητάει τον λόγο. Κύριε Χουανγκόγκ, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση η οποία μόλις ψηφίστηκε είναι ένα άσχημο χτύπημα εις βάρος του Ευρωπαίου πολίτη το ΕΛΚ και οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι θέλουν να κάνουν το λαό της Ευρώπης να πληρώσει αυτή την κρίση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συνδέσω το όνομά μου και το όνομα της Σοσιαλιστικής και Δημοκρατικής Ομάδας στο κείμενο αυτό. Παρακαλώ να αποσύρετε την υπογραφή μου. Κύριε Γκόγκ, η δήλωσή σας θα προσαρτηθεί στα πρακτικά. Βάσει της ημερήσιας διάταξης έχουμε την έκθεση του κυρίου Κόρτες Λάστρα για τη συμμετοχή της πολιτικής σύνοχης στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της στρατηγικής 2020. Έχουμε μία μοναδική Τροπολογία, τροπολογία 9, οι άλλες έχουν αποσυρθεί. Ψηφίζουμε ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το κείμενο. Η κυρία Τόγια ζήτησε τον λόγο. Να πω ότι για την προηγούμενη έκθεση, την Χουόγκ Νόκ, δεν δούλεψε το μηχάνημά μου. Εγώ καταψήφισα φυσικά. Σα ευχαριστούμε κύριε Ατόγια. Θα καταγραφεί στα πρακτικά. Θα καλέσουμε και ένα τεχνικό έκθεση παιδιών για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Μετά την παραγραφή 1, τροπολογία 2 τη Συνομόσπονδη Ενωτική Αριστερά, ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παραγραφή 3, τροπολογία 4 τη ίδια ομάδα. ψήφι κατά, αποχές, Απορρίπτεται επίση. Παράγραφο 4, τροπολογία 3 τη ΓΚΟΕ σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απέριπτε. Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη προφορίες. Επίση και το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 5 της ΓΟΕ, ονομαστική κλίση, άρχιδη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται επίση και η τροπολογία 5. Περνάμε μετά την παράγραφο 5, τροπολογία 6 τη ΓΚΟΕ σε τρία τμήματα αυτή τη φορά κάθε φορά με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα άρχεται ψηφοφορία ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση τη ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι λήξης της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τμήμα 3 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται και το τρίτο τμήμα. Μετά την παράγραφο 7 έχουμε τροπολογία 7 της ομάδας της νομός Πονδυσιανωτικής Αριστεράς. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8 Παύλα 2 τροπολογία 1 του ΕΛΚ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτό το πρώτο τμήμα τμήμα 2 ψήφι υπέρ κατά Πρέπει να το ελέγξουμε αυτό. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία επαλήτευση για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. <clears throat> Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο εκπίπτει λοιπόν. Ψηφίζουμε την παράγραφο 9 του αρχικού κειμένου. Ψήφι Κατά. Δεκτή. Παράγραφος 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 13 το κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15, αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτό. Δεύτερο τμήμα ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μετά την παράγραφο 17, τροπολογία 8, ψηφίπερ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. <clears throat> Παράγραφος 20, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται επίσης. Μετά την παράγραφο 20, τροπολογία 9, ψήφι κατά, αποχές απολύπτεται. Τελική ψηφοφορία, το κείμενο όπως τροποποιήθηκε, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται η έκθεση. Ερχόμαστε στην έκθεση Κύριλοφ για την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον Στο Νότιο Κάφκασο, παράγραφος 8, έχουμε δύο τροπολογίες. Τροπολογία 1, ψηφιπέρ <clears throat> κατά, αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, αρχιτεί ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. <clears throat> Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Παράφρος 13. Τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 14. Τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 15, τροπολογία 7, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Παράγραφος 23, τροπολογία 5, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 54, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται το συνολικό κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί ψήφι υπέρ κατά άποχες δεκτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ τα μάλα για τη συνεργασία σας. Είναι η πρώτη φορά που προεδρεύω σε, σε ψηφοφορίες. Όσοι θέλουν να φάνε, σας παρακαλώ να φύγετε ηρέμος και ησύχως, διότι πρέπει να κάνουμε και τις επεξηγήσεις ψήφου. Έκθεση Γκρέχ, ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ χαίρομαι για το ότι ψηφίσαμε μια έκθεση για τη δημιουργία